Ladies and gentlemen, please be seated. We start. Κυρίε και κύριοι, καθίστε. Θα ξεκινήσουμε αυτή την μακροσκελή αλλά και ενδιαφέρουσα διήμερη συνάντηση στην Υποβιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Ας ξεκινήσω αρχικά με την έγκριση της σημερινής διάταξης. Εάν Εφόσον δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρώ ότι έχει εγκριθεί. Να υπενθυμίσω ότι υπήρξε μία τροποποίηση στη μέση διάταξη, στο σημείο 4. Η εφαρμογή των συμφωνιών του Μίτσκ και ανταλλαγή απόψεων με την αυτοκροχότητα πρέσβη κύριο Γελισιέιεφ της Ουκρανίας και τον εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Το πέμπτο σημείο θα είναι η ενημέρωση σε ό,τι αφορά την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Κοινοβουλευτική Ολομέλεια Σύνοδο του ΝΑΤΟ και την Ερηνή Σύνοδο στη Βουδαπέστη. Εάν συμφωνείτε κι εσείς, θεωρώ εγκριθήσα την μέσα διάταξη. Να σας υπενθυμίσω ότι αναμεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίαση αυτή και για το γλωσσικό καθεστώς προτεραιότητα έχει δοθεί σε ό,τι αφορά την ερμηνεία στις γλώσσες των ε, πλήρων μελών της υποεπιτροπής μας. αν συμφωνείτε και εσείς μέλη, να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16 Απριλίου και της 6 Μαΐου. Για τυχόν παρατηρήσεις έχετε προθεσμία μέχρι σήμερα το απόγευμα. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, θα θεωρήσω ότι έχουν εγκριθεί και τα πρακτικά. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Ας περάσουμε στο σημείο 4 και πάλι να καλωσορίσουμε τον ε, πρέσβη Γελισέιεφ και το διοικητή εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, υπεύθυνο και αρμόδιο για τη Ρωσία, τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, την περιφερειακή συνεργασία και τι άλλο. Ελπίζω να τα θυμηθήκα όλα, εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Να συνεχίσω. Α, συγγνώμη, διακόπτη η Πρόεδρος. Λυπάμαι πολύ. Ε, ξέχασα να αναφέρω ότι η συνάντηση αυτή γίνεται σε συνεργασία με την Αντιπροσωπή Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία και ο κύριος Αντρέι Πλένκοβιτς, επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, βρίσκεται εδώ μαζί μας και σίγουρα θα του δώσουμε το λόγο στη συνέχεια. Αντρέι, όμως, αν μου επιτρέπεις, να δώσουμε πρώτα το λόγο ε, στον πρέσβη. Θα είστε τρίτος κατά σειρά, αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ κυρία Φωτίγκα. Αντρέη και σένα σε ευχαριστώ που μου δίνεις το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φωτίγκα και τον κύριο Πλένκοβιτς για τη διοργάνωση αυτής της επίκαιρη συζήτησης, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να καταγράψουμε και να δούμε τι ακριβώς έχει εφαρμοστεί σε διαφορά τις συμφωνίες του Μίνσκ και να διαρευνήσουμε τυχόν περαιτέρω μέτρα που μπορούν να υιοθετηθούν για την Ευρώπη. Αγαπητοί φίλοι, η Ουκρανία θεωρεί ότι οι συμφωνίες Μίνσκ είναι ο μοναδικός ε, δρόμος ε, μοναδικό δρόμο είναι η τήρηση των διατάξεων. Θέλουμε να αντικοποιήσουμε αυτό το διάλογο για την ελευθερική διαδικασία και προβλέπουμε στην ίδια βούληση και από την ρωσική πλευρά. Παρά το γεγονό ότι η ανακοχή παραβιάζεται καθημερινά, εμεί οι Ουκρανοί πληρούμε τις προϋποθέσεις για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στο έδαφος. Ξεκινήσαμε με την υλοποίηση των πολιτικών διατάξεων της Συμφωνίας του Μίνσκ, συνταγματική μεταρρύθμιση και αποκέντρωση είναι καθοδόν. Έχει ξεκινήσει το, έχουν ξεκινήσει εργασίες στις υποεπιτροπές για συγκεκριμένες ενέργειες, κοινωνική και πολιτική αποκατάσταση, αποκατάσταση ε, και ανθρωπιστική βοήθεια. Οι νόμοι για την αμνηστία και ειδικό καθεστώ για ορισμένε περιφέρειε στην Τόνμπα έχουν ήδη υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο μα. Δίνεται η εντύπωση ότι οι συμφωνίε του Μίνσκ υλοποιούνται όπως πρέπει. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει. Δυστυχώς η Ρωσία ε, και αυτοί οι εγκληματίες που στηρίζονται από τη Ρωσία ε, δείχνουν απόλυτη άγνοια, ακολουθούν τη γνωστή τακτική του σαλαμιού για να κατακαιρματίσουν, αν θέλετε, τις περιοχές και να λάβουν νέες υποχωρήσεις από την Ουκρανία και εδαφικές και πολιτικές. Αντί να τηρήσουν αυστηρά την εκεχηρία, η Ρωσία προτίθεται να κλιμακώσει τη σύγκρουση. Από τις 15 Φεβρουαρίου τρέχοντος, οι θέσεις ε, της Ουκρανίας έχουν δεχθεί ε, πάνω από 5.000 επιθέσεις και με απαγορευμένα όπλα. 108 Ουκρανοί ε, στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και 519 έχουν τραυματιστεί. Πρόσφατες επιθέσεις σε ουκρανικές θέσεις στην ε, περιφέρεια Ντανέτσκα αφορούσαν περίπου χίλιους ε, ε, μαχητές της ρωσικής πλευράς. Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε νέες ανησυχητικές εκθέσεις ό,τι αφορά την συγκέντρωση μαχητών και πολεμοθοδίων σε ορισμένες περιοχές έχουμε και ομοιρίες και παράνομες κρατήσεις. 319 Ουκρανοί εξωματούχοι παραμένουν ε, ε, κρατούμενοι, καθώς και πάνω από 40 πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι κρατούνται παρανόμως στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης και της Νάντια Σάσνικα αντί για την απόσυρση όλων των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από την Ουκρανική επικράτεια, η Ρωσία ποτέ δεν έχει σταματήσει την χρήση βαρέως οπλισμού. 42.000 ε, στρατιώτες υπάρχουν στην περιοχή και 9.000 κανονικές στρατιωτικές ε, δυνάμεις, πάνω από 500 τάγκς. πολεμικά συστήματα, συστήματα εκτόξευσης ε, πυράβλων και ούτω καθεξής. Αντί να γίνει μία συζήτηση, ένας διάλογος, ε, η Ρωσία προσπαθεί ε, να εκτροχιαστεί η πολιτική διαδικασία. Η αποστολή ε, δεν έγινε δεκτό το αίτημα να ε, επισκεφθεί ορισμένες περιοχές για να παρακολουθήσει τις τοπικέ εκλογές. Η Ρωσία αγνοεί τι δεσμεύσει τη για συγκεκριμένου μηχανισμούς για την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ρωσία έχει ήδη στείλει 28 ανθρωπιστικά κομβόι, όπως τα ονομάζει, στην Τόνβατσκ Θέλουμε την αποκατάσταση πλήρους ελέγχου στα σύνορα, κάτι το οποίο είναι ε, κρίσιμη σημασία για να σταματήσουν οι ροές ε, ε, στρατιωτικών δυνάμεων και όπλων. Όμως δεν δέχεται παρατηρητές η Ρωσία σε όλα τα συνοριακά φυλάκια. Μια περιοχή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός του ελέγχου της Ουκρανίας. Θέλουμε να να σταματήσουν οι αποστάσεις αποσταθεροποίησης ε, της κατάστασης στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις πολύ συχνά φτάνουν στην επικράτειά μας και διενεργούν τις εγκληματικές τους ενέργειες και για τις ε, περιοχές της Περνιστερίας υπάρχουν ζητήματα και έτσι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο όλου αυτού του διαδρόμου των 700 χιλιόμετρων. Γι' αυτό και στοχεύει την αποσταθεροποίηση της κατάστασης σε ορισμένες πόλεις της Ουκρανίας και προτιμά αυτή τη δίωδο. Οδυσσός, Μαριανούπολη και ούτε καθεξής. Μάλιστα, οι ε, τακτικές στρατικές δυνάμεις της ε, Ρωσίας τρομοκρατούν τους αμάχους και με την καταστροφή κρίσιμης ε, υποδομής. Την περασμένη εβδομάδα ε, κατέστρεψαν έναν αγωγό στον Ντονέτσκ και έτσι πάνω από μισό εκατομμύριο πολιτών δεν είχαν φυσικό αέριο για πολλές ημέρες. Ο ρόλος του Κρεμλίνου είναι κατανοητός και γνωστός. Θέλει να διαταράξει τη διαδικασία του Μίνσκ με το να ασκεί πιέσει στην ε, Ουκρανία. Εμείς με τα βίας ε, καταφέρνουμε να ε, διατηρούμε στη ζωή την ενεργητική διαδικασία, ε, γιατί δείχνουμε μετριοπάθεια και αυτοσυγκράτηση. Όμως αυτό δεν επαρκεί για την επαναφορά της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Απλώς έχει στόχο να μειωθούν τα θύματα από την πλευρά Ουκρανίας. δεν θα πρέπει να πιστέψουμε τα προπετάσματα καπνού της ε, Ρωσίας, γιατί οι δεσμεύσεις πρέπει να μεταφραστούν σε πραγματικές και απτές πράξεις. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τίποτα σοβαρό δεν συμβαίνει στην ε, Ανατολική Ουκρανία, εφόσον ε, έχει μειωθεί ο αριθμός των μαχών. Γιατί υπάρχει έλλειψη νομοθετικής ε, δράσης σε αυτό το στάδιο που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ε, στη συνολική αιστεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα είναι πιο δύσκολο να καταπολεμηθεί και να κατασβεστεί η πυρκαγιά. Πολλές φορές σας έχω πει, φίλοι μου, ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε πέντε βασικούς πυλώνες. Πρώτον, να ενισχύσουμε την ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία. Δεύτερον, οικοδόμηση διατλαντικής αλληλεγγύης. Τρίτον, περισσότερες διπλωματικές προσπάθειες και άσκηση πιέσεων στη Ρωσία. Τέταρτον, να επενδύσουμε σε, στο success story της Ουκρανίας και τέλος να παροτρύνουμε τη Ρωσία να αποκαταστήσει το, ένα κράτος διεθνούς δικαίου ε, με την εισαγωγή νέων περιοριστικών μέτρων επειδή υπάρχει υψηλό αριθμό προκλήσεων, έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε σοβαρά το ενδεχόμενο εισαγωγή νέων κυρώσεων, ούτω ώστε να αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Ε, ε, οι ε, επιθέσει στη Μαριούπολη δεν μπορούν να θεωρηθούν αφορμή, έναυσμα. Πρέπει να τι αποτρέψουμε και όχι να, δώσουμε νέες, να κάνουμε νέε επιθέσει. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε νέε επιθέσει για να, για να εισάγουμε νέα μέτρα περιορισμού της Ρωσίας, όπως έγινε ε, με την κατάρριψη του MA17. Πρέπει να υπάρξει έγκαιρη και αποφασιστική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς οι μετριοπαθείς αντιδράσεις από τους θύτες ε, θα θεωρηθεί απλή δηλία ε, και έτσι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν συνάδελφοι να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για να στηρίξουμε την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο λεγόμενο soft power της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει εμείς να παρουσιάσουμε μια εναλλακτική στην έννοια του Ρουσκιμίρ ε, για να κερδίσουμε το πνεύμα και την καρδιά των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Ε, πρώτον, ε, ε, απαλλαγή από τις θεωρήσεις. Προστασία των πολιτών στην Ανατολική και Κεντρική Ουκρανία. Καταπολέμηση της ρωσικής προπαγάνδας. Και τέταρτον, να δώσουμε μια ε, ευρωπαϊκή προοπτική στα πιο φιλόδοξα τμήματα και χώρε τη ε, Ανατολική Τερική Σχέση. Τώρα, να περάσω στο λεγόμενο hard power τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω σε ό,τι αφορά την ε, ΚΕΠΑ, η οποία μπορεί να αφορά, να αφορά για παράδειγμα, τα εξή βήματα. Να δώσουμε αρχικά στην Ουκρανία δεδομένα του δορυφορικού κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούσαμε να έχουμε έτσι επίβλεψη και των συνόρων με τη Ρωσία. Να ενισχύσουμε την εντολή της ε, Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, αποστολή της κοινή ε, πολιτικής άμυνας να ξεκινήσει όπως έχει προτείνει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία CSDP δεν έρχεται σε αντίθεση με την Συμφωνία Μίνσκ, αλλά θέλει να την ενισχύσει. Δεν θα αντικαταστήσει την αρμοδιότητα του ΟΗΣΥ, αλλά συμπληρώνει τη δράση του επιτόπου. Θα επικεντρωθεί στι ε, πτυχε ασφαλεία αυτή τη κατάσταση για να αποτρέψουμε περαιτέρω επιδείνωση. Πρέπει να ε, συμπληρωθεί το κενό της ασφάλειας και αυτή τη μεταβατική περίοδο σε αυτήν την περιοχή. Πολλοί θα συμφωνήσετε ότι η εντολή της αποστολής OECM είναι ιδιαίτερα στενή για να διασφαλίσει την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ και κυρίως επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της εκεχηρίας και της επαλήθευσης της απόσυρσης των όπλων. Πολλές όμως πτυχές της ειρηνευτικής διαδικασίας δεν έχουν εφαρμοστεί. Γι' αυτό θα αναφέρω μόνο συγκεκριμένε περιπτώσεις όπου η Ουκρανία χρειάζεται επιγόντως περαιτέρω βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εμπειρία της Ένωσης στην επίλυση διαφορών και συγκρούσεων. Πρώτον, ε, κατάρτιση των νομικών μας υπηρεσιών για να αποτρέψουμε περαιτέρω ενέργειες της ρωσικής πλευράς. Κατάρτιση των, της επωνομαζόμενης ε, πολιτοφυλακής ε, της τοπικής Ε, ανοικοδόμηση και αποκατάσταση των περιοχών κατόπιν των συγκρούσεων που έχουν επιστρέψει δηλαδή στην επικράτηση της Ουκρανίας μετά δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους παρατηρητές και πυρογνώμονες του ΟΗΣΥ που θα ε, προετοιμάσουν και θα παρακολουθήσουν τις τοπικές εκλογές. Άλλο ένα πιεστικό ζήτημα είναι η παροχή ανθρωπιστικής συνδρομής στις κατεχόμενες περιοχές. Και τέλος, κοινή δήλωση της 12 Φεβρουαρίου. Γαλλία και Γερμανία δεσμεύτηκαν να παράσχουν τεχνική συνδρομή για την αποκατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην Donbass με τη θέσπιση διεθνούς μηχανισμού για την Εκταμείευση κοινωνικών επιδομάτων. Πώς θα διασφαλίσουμε όμως την εφαρμογή αυτής της δέσμευσης. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιηθούν υπό την ομπρέλα αυτή. Όπως γνωρίζετε, τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Αποστολή επισκέφθηκε την Ουκρανία για να εξετάσει τις ιδέες της Ουκρανίας. Ήταν μια καλή αρχή, αλλά αυτή τη στιγμή ε, δεν υπάρχει κάποια συνέχεια. Γι' αυτό, συνάδελφοι, να επενθυμίσω ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού για τη χρηματοδότηση της κοινή ε, πολιτικής ε, άμυνας και ασφάλειας του Μαΐου, που εντοπίζει και αναφέρει ότι είναι πολύ μικρή η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία. Και στηρίζω και άλλο ένα σημαντικό πόρισμα τη έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερα μέσα και δυνατότητες μόχλευσης από οποιοδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό για την επίλυση της σύγκρουση. Στην πολιτική, η πολιτική ασφάλειας και προστασίας μπορεί να συμπληρωθεί και με άλλα μέσα και μηχανισμούς χρηματοδοτικούς. Γι' αυτό είναι κρίσιμη σημασία να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην κατάσταση στην Ουκρανία θα συμβαδίζει με το ρόλο που μπορεί να δραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση κρίσεων και συγκρούσεων. Μία ισχυρή ανταπόκριση και αντίδραση στην επιθετικότητα της Ρωσίας είναι βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Επίσης, προορατική ε, επένδυση στο success story της Ουκρανίας θα είναι βασικός ε, ε, κινητήριος δύναμη ε, για την αλλαγή στην ευρύτερη περιοχή. Και τέλος, ε, η διασφάλιση της σωστής διενέργειας της ειρηνευτικής διαδικασίας. Για να γίνει μάλλον όλο αυτό, πρέπει να βολιδοσκοπήσουμε το τι συμβαίνει επί τόπου, να δούμε ακριβώς τι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό ευχαριστώ και τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές που επισκέφθηκαν αυτές τις περιοχές και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει και μία αποστολή πρέσβεων στην περιοχή. Και είπα ότι εκπρόσωπος, κυρία Μογκερίνη, επίση θα επισκεφθεί τη χώρα μου ε, ή θα ήθελε να επισκεφθεί τη χώρα μου για να καταγράψει τα όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους 7 μήνες που έχουν περάσει από την περασμένη της επίσκεψη. Σας ευχαριστώ. Thank you, Ambassador. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Επόμενο αγορητή. Ευχαριστώ. Μετά από αυτά τα σαφή και ξεκάθαρα λόγια του Πρέσβη, ε, με τον οποίο είμαστε πενήθηκα εδώ και χρόνια και εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία του. Ο τίτλος της συνεδρίας είναι «Εφαρμογή των ε, συμφωνιών». Φυσικά αυτό δεν αφορά πρωτίστως την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσους συμμετείχαν στις συμφωνίες αυτές και στη σύναψή τους. Θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω, σύμφωνα με το πνεύμα το οποίο μίλησε και ο πρέσβης, για την πρόσφατη επίσκεψη στην Μαριούπολη, αλλά και σε άλλες πόλεις που έχουν εμπλακεί στην σύγκρουση. Αύριο με τον Επίτροπο Χάν θα μεταβούμε στην Ουκρανία να, να συναντήσουμε τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον Πρόεδρο της Βουλής αλλά θα πάμε να δούμε και τα προγράμματα που στηρίζει η Ένωση στην περιοχή. Τώρα, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνίων του ΜΙΣΚ, να σας υπενθυμίσω αυτά που αποφάσισαν οι αρχικοί κρατών το Μάρτιο. Μόλις δηλαδή πριν από τρεις μήνες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από όλους, όλα τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως τις συμφωνίες του Μίνσκ ε, τονίζοντας την ευθύνη της ρωσικής πλευράς και δήλωσε ότι η Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει τις συμφωνίες αλλά και να τις ε, ελέγξει κατά την εφαρμογή τους και να συνεχίσει τις προσπάθειες σε ε, ζητήματα CFDA και ενεργειακής φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει λοιπόν την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Δύο από τα μέλη της έχουν συμμετάσχει στις σκληρές διαπραγματεύσεις. Η στήριξη της ειδική αποστολής έχει κοστίσει μέχρι τώρα 25 εκατομμύρια ευρώ και προς το παρόν υπάρχουν 500 άτομα τα οποία εργάζονται για αυτές τις συμφωνίες και προβλέπουμε να ανέρθουν σε χίλιους Υπάρχει λοιπόν και παρακολούθηση των, της και με τεχνικά μέσα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε χορηγήσει 64 οχήματα, ε, από των οποίων τα μισά είναι ε, εξοπλισμένα. Τα τρία θέατα του προσωπικού της αποστολής είναι ε, ε, πολίτε τη Ένωση, καθώς επίση και η χρηματοδότηση κατά τρία τέταρτα πρόκειται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίες λοιπόν του ΜΙΣΚ θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και τώρα θα σα μιλήσω για την κατάσταση που επικρατεί, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι το οποίο τόνισε, τόνισαν οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων, ότι δηλαδή η διαδικασία που έχει εφαρμοστεί στα ενεργειακά ζητήματα έχει αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα και ε, σύντομα θα υπόγραφει από τους υπουργούς Ουκρανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Ο αντιπρόεδρος Εύκοβιτς επίσης θα υπογράψει τη συμφωνία και θα διεξαχθεί και το διατησία της στο Στοχόλμης τον Ιούλιο όπως ξέρετε συζητήσεις για το CFTA η εφαρμογή συνεχίζεται, είναι σαφές και αυτό έχει καταστεί σαφές στην διάσκεψη της Ουκρανίας και αναζητούμε τρόπους για να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία η οποία παρέχει η συμφωνία για την ε, ικανοποίηση και των ε, εμπλεκομένων πλευρών. Τώρα, η εφαρμογή της συμφωνίας του ΜΙΣΚ, η κατάσταση στην δομή της ασφάλειας ε, έχει βελτιωθεί από την κατάψη του του Φεβρουαρίου πέραν των τραγικών γεγονότων που έγιναν στην αρχή. Συνεχίστηκαν εντάξει, οι συγκρούσεις και πολλά και πολλές ε, συγκρούσεις έγιναν στην περιοχή του Ντόνιεσκ και στο Ντούκασκ. Αυτό σημαίνει ότι κεντρικά και νότια ε, συνεχίζονται οι συγκρούσεις. Ε, φυσικά αυτό είναι αποτελεί στοιχείο ανησυχίας και το πρόσφατο γεγονός ήταν αυτό το οποίο Αναφέρθηκε και ο πρέσβης και που θεωρήθηκε από τον από εμά ως, ως παράβαση της κατάψης του πυρός από τότε που συνήθισε η συμφωνία του Μίνσκ και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη σύγκρουση βαρέα όπλα. Αυτό το συμβάν λοιπόν ήταν σημαντικό αλλά δεν ήταν το μοναδικό που μας ανησύχησε ικανός αριθμός βαρέων όπλων έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα και κυκλοφορούν. Αυτό το αναφέρει η αποστολή του, του που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή. Υπάρχει και συνεργασία με την Κοινή Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία συμμετέχουν ε, αξιωματούχοι της, Ρωσία Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση δεν είναι διόλου απλή. Ο πρέσβης αναφέρθηκε στην ε, απελευθέρωση ομήρων 319 Ουκρανοί στρατιώτες κρατούνται παρανόμως. Η πολιτική διαδικασία και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην εργασία του Χέντι Τελιαβίνη της οποίας η εντολή Πάβη το τέλειο του μήνους έκανε σκληρή δουλειά κάτω από, από συνθήκες περίπλοκες και δύσκολες. Μέχρι τώρα δεν έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα ζητήματα τα οποία θέτουν τα άτομα που επιθυμούν την απόσχηση αφορούν το θέμα των διεξαγωγής εκλογών έχει η ο ECD έχει συντάξει μια έκθεση και έχει ζητήσει από τον πρέσβη Λούκας να κάνει τις απαραίτητες προπαρασκευές. Διότι όπως καταλαβαίνει θα πρέπει να υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την διεξαγωγή των εκλογών. Αυτές οι τοπικές εκλογές θα διεξαχθούν είτε σύμφωνα με τις συνολικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ουκρανία είτε τις τοπικές που διεξαχθούν στην περιοχή. Θα πρέπει όμως οι προϋποθέσεις να υπάρχουν προηγουμένως πριν την κήρυξη των εκλογών. Επιπροσθέτως και άλλα θέματα έχουν σημασία πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών σε ανθρωπιστική βοήθεια η οποία θα προέρχεται όχι μόνο από ρωσικής πλευράς αλλά και από άλλες πλευρές. Ο πρέσβης αναφέρθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να πω ότι αυτοί οι δεσμοί θα πρέπει να αποκατασταθούν. Υπάρχουν Γερμανοί και Γάλλοι εμπειρογνώμονες που εργάζονται, αλλά δίχως εγγύηση ασφάλειας δεν μπορεί να επιτευχθεί. Το επόμενο θέμα είναι να αποσυρθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις και να αφοπλιστούν οι παράνομες οργανώσεις και να δεξαχθούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Θα ήθελα εδώ να σχολιάσω αυτό το είπε ο πρέσβης. Πρόκειται για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που θα ε, διασφαλίζουν αυτό το καθεστώς ειδικά με το Λουγκάνσκ που θα πρέπει να αντανακλάται στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και πρέπει να ψηφιστεί φέτος κατά τη δεύτερη ανάγνωση αλλά και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα πιέζουν. Τέλος, χρειάζεται να αποκρισταθεί ο Ουκρανικός έλεγχος των συνόρων με τη Ρωσία μέχρι τα τέλη του έτους. Αυτό είναι ένα ζήτημα απαραίτητο διότι αυτή τη στιγμή τα σύνορα δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ουκρανικών αρχών αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί σύμφωνα με τη Συμφωνία του ΜΙΣΚ όταν ε, πραγματοποιηθεί η συνταγματική μεταρρύθμιση. Όλες αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να οδηγήσουν στο να καταστήσουν αυτές τις προϋποθέσεις πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενικά Διευθυντά. Ο κύριος Πλένκοβιτς τώρα από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία την διακοινοβουλευτική με την Ουκρανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φωτίγκα, αγαπητέ πρέσβη, αγαπητέ διευθυντή, αγαπητοί συνάδελφοι. Πάντα είναι καλό και ωφέλιμο να υπάρχει τέτοια συνεργασία με την Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει το θέμα αυτό στην ε, ημερήσια διάταξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ, βασικό θέμα για την ε, ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ειρηνική ε, επίλυση της διαμάχης να τονίσω ότι καταρχάς τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κύριος Βίγκαν, ο πρεσβευτής σε ό,τι αφορά τα 13 μέσα τα οποία περιλαμβάνονται στη συμφωνία του Μίντς και γιατί είναι τόσο χρήσιμη η εφαρμογή τους. Η δυναμική της εφαρμογής και η χρονική συγκυρία δεν ήταν απόλυτα ικανοποιητική. Αυτό εξαγάγουμε συμπέρασμα επειδή πάνω από 100 Ουκρανοί στρατιώτες ε, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Και φυσικά η ανταλλαγή ομήρων, η απόσυρση όλων των δυνάμεων ήταν ένα θέμα. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύω ότι η έκκληση της Ουκρανικής κυβέρνησης και του Προέδρου για μεγαλύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή στη διάσταση της ε, άμυνας και της ασφάλειας που αποτελεί και αρμοδιότητα της Επιτροπής μας είναι σημαντική. Στο Συμβούλιο, εξ όσων ακούω, γίνονται διαβουλεύσεις για το πώς θα ενισχυθεί η συμβουλευτική αποστόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάφοροι εξημών έχουμε επισκεφτεί το Κίεβο και ο ρόλος της αποστολής έχει σημαντική είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την προστασία των αμάχων. Χρειάζεται λοιπόν, ε, μάλλον θα εκτιμούταν ιδιαίτερα από πλευρά τη Ουκρανία μεγαλύτερη δέσμευση. Κάτι άλλο που πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δηλωθεί στην παρούσα φάση είναι το εξή. Δεν μας απασχολεί μόνο τον Ντόμπας. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χάσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία όταν συζητάμε την, ε, το θέμα της Ουκρανίας για να αναφέρουμε την Κρυμαία που έχει προσαρτηθεί παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι απαράδεκτο και πάντα δηλώνεται ξεκάθαρα στα, στις δηλώσεις και τις διακηρύξεις και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να γίνεται αναφορά στην ε, διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης, γιατί αυτό αποτελεί ένα τμήμα τη ευρύτερη συμφωνία του Μίνσκ. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι διεθνεί οργανισμοί θα έπρεπε να υποστηρίξουν το έργο διευκόλυνση, όπω ε, είπε η κυρία Ταλιαντίνη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρξει κάποιο είδου επικοινωνία και κάποια στοιχειώδη ε, ε, εμπιστοσύνη με την άλλη πλευρά του μετώπου. Αυτό είναι φυσικά πολύ περίπλοκο, πολύ ευαίσθητο θέμα αλλά αυτό καταδεικνύει η εμπειρία και κάποιων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι με τα διάφορα μέτρα από η αμνηστία, χορηγήση εγγράφων, πρόνοια για τους πρόσφυγες. Όλα αυτά είναι χρήσιμα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον τόμα μας. Τώρα, μια πιο καινοτομική προσέγγιση. Όσο περνάει ο καιρός νομίζω θα χρειαζόμαστε μια διεθνώς ορισμένη προσωπικότητα που θα αναλάβει τη διευκόλυνση και την πρόθεση της κατάστασης. Αυτό πιστεύω ότι είναι μια ιδέα που θα, ιδέα που θα μπορούσε να βοηθήσει την Ουκρανία και να βελτιώσει τα αποτελέσματα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με... Βρέθηκα λοιπόν, παρευρέθηκα στο Κίεβο στις 3 και 4 Ιουνίου όταν έγινε η επίθεση στο Μαρίνκα και θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήταν αυτό λίγο πριν την ομιλία του Πρόεδρου Πολοσέγκο την επόμενη μέρα για την κατάσταση της Ένωσης. Δεν ήταν λοιπόν τυχαία η χρονική συγκυρία, ασφαλώς. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ε, στην περαιτέρω διαμόρφωση των πολιτικών μας και χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ και διάφορα μέλη της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Άντρα, και τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε τη συζήτηση, επιτρέψτε μου να εκφράσω μία παρατηρήση. αν θα μπορούσε ο κύριο Βίγκαν στις απαντήσει να μας περιγράψει το πώ προχωράει η ομάδα επαφή του Μίνσκ. Γιατί είναι λίγο αντιφατικά τα αποτελέσματα που ακούμε από την τελευταία συνάντηση. Η Ουκρανική πλευρά κηρύσσει την ρήξη των διαδικασιών από τη ρωσική πλευρά, ενώ ο πρέσβης Χαντιντελαβίνη ήταν μάλλον ουδέτερος, μάλλον ουδέτερη. Δήλωσε ότι είχε αποφασιστεί η επόμενη συνάντηση, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία της συνάντησης. Προκλήθηκε λοιπόν Μια σύγχυση. Θα προτιμούσα προσωπικά ε, πιο ενεργό ρόλο των διπλωματών που συμμετέχουν στην ε, αποστολή του ΑΣΕ. Τώρα όμως ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κατά αρχάς ο κύριος Κέλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Οι συμφωνίες του Μίνσκ δεν ε, έχουν εφαρμοστεί. Το θέμα είναι σε τι βαθμό εξακολουθούν να ισχύουν αλλά εκ παραλίλου πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι το μοναδικό πλαίσιο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μα. Άρα είναι προ το κοινό μα συμφέρον να ενισχύσουμε τη συμφωνία αυτή. Ο στόχο δε του να ε, εφαρμοστούν πλήρους είναι κοινό στόχο. Ο Ουκρανό πρέσβη μα παρουσίασε εντυπωσιακά περιστατικά. Εκατοντάδες ε, νεκροί, πάνω από 300 φυλακισμένοι και η Νάτια Το βασικό νομίζω για μας είναι να μην ε, συνηθίσουμε σε αυτή την επανάληψη των παραβιάσεων. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε, κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και σοβαρό. Η δε βάση για τις δράσεις μας είναι το ψήφισμα της περασμένης εβδομάδας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας που προετοίμασε και κατήρτησε ο συνάδελφος Λαντσμπέργκης και βασίζεται σε μια αυστηρή ρεσιμότητα. Καταρχάς, η Ρωσία θα πρέπει να συμφωνήσει με τη συμφωνία του Μίνσκ και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πρώτα βήματα για κάποια ομαλοποίηση των σχέσεων. Αυτό ασφαλώς συνεπάγεται ότι οι κυρώσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να συνεχίσουν και θα πρέπει μάλιστα να ενισχυθούν καθότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική σε ό,τι αφορά τις διαρκείς παραβιάσεις της ε, συμφωνίας του Μίνσκ. Έχουμε λοιπόν πολύ πιστικά σήματα που μας καταδεικνύουν ότι λειτουργούν οι κυρώσεις και ότι η ρωσική ηγεσία ε, είναι σε σημείο απελπιστικό σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Είναι λοιπόν το θέμα κατά πόσο θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε ενότητα και αποφασιστικότητα να τα συνεχίσουμε τα μέτρα αυτά. Στη συνέχεια, κάτι άλλο πολύ σημαντικό, από ό,τι φαίνεται από την παρουσίαση και των δύο ε, πρεσβευτών, είναι ο έλεγχος των στα ουκρανικά σύνορα. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ευκαιρίες ε, εγγυήσεις προκειμένου οι παρατηρητές να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά του σύμφωνα με την Συμφωνία του Μίνσκ. Στη συνέχεια, ο πρέσβης ε, μίλησε για τη ρωσική θεωρία η οποία δεν έχει ε, εξεταστεί με τον πρέπον τρόπο, με τον ε, δέοντα τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την θεωρητική βάση για την ε, Ουκρανική εισβολή για να προασπιστεί μόνο μερός τους συμπατριώτες ε, εκτός ε, Ρωσίας χρησιμοποιώντας στρατιωτική δύναμη. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ουκρανία, ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Καθότι Κάθε χώρα θα μπορούσε να μπει στο στόχαστρο στην περίπτωση αυτή με τη δικαιολογία τη ε, υπεράσπιση, προάσπιση των συμπατριωτών Ρώσων στην Αλαδαπή. Το δικαίωμα στρατιώτική παρέμβαση, δηλαδή στις, ε, στα ιστορικά άλλες χώρες, Να σα υπενθυμίσω τον Πρωθυπουργό Λάμπαροθ στο Μόναχο φέτος, ο οποίος και δήλωσε ότι Η Ουκρανική κρίση θα πρέπει να θεωρηθεί εργαλείο άσκησης πίεσης στις δυτικές δυνάμεις, προκειμένου να συμφωνήσουν για μια νέα διεθνή σταθερότητα, ένα νέο σύστημα διεθνούς σταθερότητας, το οποίο ερμηνεύει τους, ε, τις κινήσεις της Ρωσίας το σύμφωνο και το πρότυπο Μολόφ Ρίμπετρον. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο πρέσβης, να προβλέψουμε εν το χρόνο και εγκαίρως ε, την συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία μαζί με άλλες ε, βασικές ε, μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Και ο επόμενο είναι ο κύριος Πρώην. Παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Ναι, θα είμαι σύντομο ως συνήθω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δυο λόγια και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρέσβη κύριο Γελισέηφ για την ε, στεναρή του θέση. Νομίζω ότι η κρονική κυβέρνηση μπορεί να είναι υπερήφανη που έχει ένα τέτοιο εκπρόσωπο σε μια τόσο σημαντική θέση. Και πάλι άκουσα τα όσα είπατε και κάπως ε, χάθηκα με όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε ότι ακόμα λείπουν στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ. Από την άλλη, αρκετά στοιχεία δεν αναφέρθηκαν που πολύ συχνά αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. ως ε, τομείς αλλαγής πολιτικής στην Ουκρανία, που είναι εξαιρετικά σημαντικά και προσφυλή για μας θέματα. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση της διαφθοράς που σοβεί στη χώρα σας. Ακόμα πρέπει να ε, επανεξετάσετε ένα σύνταγμα αυτό το Σύνταγμα να περιορίσετε την εξουσία των ολιγαρχών που έχει ε, διαβρώσει, αν θέλετε, ε, τις ε, πλουτοπαραγωγικές σας πηγές ή η αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουκρανία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημεία που πρέπει να εφαρμοστούν και να βελτιωθούν. Ποια είναι η θέση η δική σας και της χώρας σας σε αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ, Μαρκ Γιούρεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν εξετάσουμε τα γεγονότα των περασμένων τριών εβδομάδων, είναι σαφές ότι πρέπει να έχουμε άμεση και αποφασιστική πολιτική αντίδραση εάν υπάρξει κλιμάκωση της ρωσικής ε, επίθεσης στην Ανατολική Ουκρανία. Οι οικονομικές κυρώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο παρότι οι απόψεις διήστανται ως προς αυτό. Για παράδειγμα, η Αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι δεν επαρκούν τα μέτρα αυτά. Οι Ουκρανικές αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι δικές μας αντιδράσεις για να επαναφέρουμε την ευρύτερη περιοχή σε μια ισορροπία, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να μην συμβεί, να την αποτρέψουμε αυτή την επίθεση της Ρωσίας δεν είναι πάντα ωραίο να είναι κανείς να έχει πάντα δίκιο, αλλά να επενθυμίσω ότι στο παρελθόν στο Κοινοβούλιο δεν θέλαμε ε, να ακούσουμε τον πρόεδρο προσέγγιση και να στείλουμε άλλες ε, δυνάμεις στρατιωτικές, αστυνομικές ή άλλες προς την Ουκρανία. Που αυτή η έκκληση ακούστηκε πριν από δύο εβδομάδες και άκουσα την απάντηση ότι η Επιτροπή δεν θέλει να το χειριστεί αυτό το ζήτημα. Εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να λάβουμε θέση. Θα έπρεπε να είχαμε στηρίξει εδώ και πολύ καιρό αυτή την έκκληση του Προέδρου. Άλλο θέμα τώρα. Ποια θα είναι η δική μας αντίδραση, ποιο είναι το κύριο σημείο σε ό,τι αφορά την ε, Ρωσία. Η επιτάχυνση της προσχώρησης της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, η ενίσχυση της άμυνας των ε, ε, πλέον ευάλωτων ε, χωρών Λετωνία, Λετωνία-Εσθονία. Πολλές φορές ακούω επικρίσεις ότι υπάρχει ανταγωνισμός ότι αφορά τα γεωπολιτικά και το καθεξής. Όχι, είναι θέμα δικής μας ασφάλειας και προστασία των εταίρων μας, όπως είναι η Ουκρανία. Εμείς, ε, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να απαιτήσουμε την ενίσχυση της άμυνας της ε, Λετωνίας και της Εστονίας. Να διεκδικήσουμε ε, μια κατάλληλη απάντηση στην έκκληση του Πρόεδρου Ποροσέγκο. Εμείς με με το να επιβάλλουμε ακόμα οικονομικές κυρώσεις σε πέντε ακόμα άτομα δεν θα επιλύσουμε το ζήτημα. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και αυτό το ζήτημα της ανατολικής εταιρική σχέσης και όλα αυτά συνδέονται και με τις εκλογές και στην Ουκρανία. Βεβαίως εμείς θέλουμε να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις Λογικό είναι να τις θέλουμε, όμως ταυτόχρονα ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Γιατί ο Πούτιν αυτό το κόλπο ε, αξιοποιεί, πιστεύει ότι όσο περνάει ο καιρός θα, θα παγιωθούν ας πούμε κατακτήσεις της Ρωσίας. Αν εμείς δεν έχουμε λοιπόν μία έτοιμη απάντηση, θα είμαστε συνυπεύθυνοι για την κλιμάκωση της ε, σύγκρουσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Στετίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μία είναι η μεγάλη μου ανησυχία ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ έχουν πεθάνει. Και να σας πω γιατί. Γι' αυτό ο κύριος Πρέσβης χρησιμοποίησε την εξορολογία soft power και hard power στο Στρασβούργο πολλά και ακούσαμε το soft power. Το hard power πρώτη φορά το ακούω σήμερα από τον πρέσβη. Ωστόσο, πιστεύω ότι η συχνότητα χρήσης αυτής της έκφρασης θα αυξηθεί. Επειδή υιοθετήσαμε δύο σημαντικά ψηφίσματα το ένα το εκπώνησε ο κύριος Πάσκου της περασμένη εβδομάδα. αυτό το ψήφισμα. Είπε λοιπόν ο κύριο Πάσκου ότι οι ενέργειε του ρωσικού στρατού είναι μια μεγάλη επίδειξη ισχύω. Και κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια αντίστοιχη επίδειξη ισχύω στην Μαύρη Θάλασσα μαζί με τις συναδελφικές δυνάμεις. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του hard power. Το soft power, κατά τη γνώμη μου, είναι κυρίως ε, η επιχειρηματολογία και ξέρουμε ότι τα ψέματα είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η ρωσική πλευρά και πάντα δείχνουν ή φαίνεται να δείχνουν ότι είναι αδύναμη η δική μας επιχειρηματολογία, το δικό μας soft power. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ρωσία σέβεται μόνο τους ισχυρούς ε, αντιπάλους. Ο πρόεδρος Ρέγκαν που κέρδισε τον ε, ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία ε, τύχανε ε, του σαβασμού της ρωσικής πλευράς. Και αν θέλουμε να μας σέβεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή η Ρωσία, πρέπει να επικεντρωθούμε στο hard power, όπως ανέφερε και ο πρέσβης. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντσμπέργκης. Okay, sorry. Εντάξει. Και κανιάτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα από την ίδια πλευρά βρισκόμαστε από ό,τι ξέρω. Είμαι πρώην διπλωμάτης. Είναι πολύ αντιδιπλωματικό αυτό που θα πω. Ναι, τσε κάνουμε επιτρέπεις και εσύ, βεβαίως. Και εγώ θεωρώ ότι το Μίνσκα έχει πεθάνει. Κατανοώ ότι δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο για μας για να γίνει αυτός ο διάλεγος και να αναζητήσουμε μια λύση, γιατί η λύση μπορεί να είναι μόνο πολιτική. Όμως, περίμενα σαφέστερη διατύπωση σε ό,τι αφορά την ε, παραβίαση της συμφωνίας του Μίνσκ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου λυπήθηκα ιδιαίτερως ε, για την καταψήφιση του ψηφίσματος ε, για τις σχέσεις ευρωπαικη Ένωσης Ρωσία και για την στρατηγική για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, ιδίω στην παράγραφο 16 που κάνει λόγο για ενίσχυση της ε, συνεργασίας για την ασφάλεια μεταξύ Ουκρανίας, Μολδαβίας και Γεωργίας και των χωρών του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή Ρουμανία και Βουλγαρία. Πολλοί με προβληματίζουν οι φήμες μετά από μια εκστρατεία που έγινε από τον Πρόεδρο Πούτιν, μάλλον την εκστρατεία γοήτρου αν θέλετε του Πρόεδρου Πούτιν στην Ιταλία και αλλού. Πρέπει να ληφθεί απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις κυρώσεις. Θα παραμείνουν μέχρι τα τέλη της χρονιάς. που είναι και η τελική προθεσμία για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εκεχηρία του Μίνσκ. Όταν η Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να παραχωρήσει πλήρη έλεγχο των συνόρων ε, με την Ουκρανία στην Ουκρανία. Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις που ε, αναφέρονται στην ε, Συμφωνία Μίνσκ 2. Εάν υπάρξει αναθεώρηση των κυρώσεων, τότε δεν υπάρχει καμία κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υφίσταται πλέον. Για χώρες όπως ε, τα κράτη της Βαλτικής, αυτό είναι ισχυρότατο μήνυμα που θα δώσει το Συμβούλιο σε μερικές ημέρες. Ευχαριστώ. Άρα, κύριε Λανσπερκής, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Δύο παρατηρήσεις για τις εκθέσεις που υιοθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Μία έκθεση ευρωπαικη Ένωσης Ρωσίας, αυτή η έκθεση μάλλον, αναφέρει μία δήλωση που καταφέραμε να ενσωματώσουμε στο τελικό κείμενο που μιλάει για τις συμφωνίες Μίνσκ όχι μόνο αναφέρει ότι οι συμφωνίε θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρω, αλλά στην αγγίλη αναφέρει και τι ακριβώ εννοούμε με αυτό. Υπήρξε ενδιαφέρουσα συζήτηση στι πολιτικέ ομάδε του Κοινοβουλίου. Γιατί χρειαζόμαστε αυτέ τι αγγίλε. Δεν είναι σαφέ τι ακριβώ εμπεριέχουν αυτέ τι συμφωνίε. Εμεί θεωρήσαμε ότι όχι, δεν είναι σαφέ. Και υπάρχει κίνδυνο που ανέφεραν ορισμένες, ε, ορισμένοι συνάδελφοι προηγουμένω. Κατά πόσο υπάρχει ακόμα ε, δυνατότητα επιτυχία των συμφωνιών Μίνσκ ή όχι, αν έχουν πεθάνει ή όχι όπως ανέφεραν. Ε, πρέπει να εφαρμοστούν πολύ συγκεκριμένα αυτά στοιχεία που είναι εύκολα να ελεγχθούν, δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα και μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε αν λειτουργούν ή όχι. Ας έχετε λοιπόν αυτά τα στοιχεία κατά νου στην παράγραφο 6 για να σας βοηθήσω. Κάτι άλλο για την επόμενη έκθεση που πολύ σωστά ανέφερε η Σάντρα, ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μικρό κύματος για την Επιτροπή Πάσχου για την κατάσταση στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Κρίμα που κάποιες από τις τροπολογίες που εγώ κατέθεσα ε, καταψηφίστηκαν. Όμως, δράτω με τις ευκαιρίες για να τις επισημάνω. Μία από αυτές ανέφερε την αυξημένη συνεργασία μεταξύ ε, Ουκρανίας, Μολδαβία και Γεωργία. σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του στρατιωτικού. Για κάποιου λόγου, οι συνάδελφοί μα στο Κοινοβούλιο θεωρούσαν ότι είναι υπερβολική η διατύπωση και την καταψήφισαν. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει ω πολιτική δήλωση. Υπήρξαν πολλά μέλη του Κοινοβουλίου, περίπου 200 μέλη του Κοινοβουλίου, που θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα καλό μήνυμα να αποστείλουμε σε αυτέ τι τρει χώρε. Ότι η αυξημένη, ενισχυμένη συνεργασία και στον στρατιωτικό τομέα είναι ένα καλό σημάδι για την ε, ενίσχυση τη ασφάλεια, αλλά και για την καλή βούληση και συνεργασία σε αυτή την περιοχή που μπορούμε να αποστείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε κύριε Φραντσουλίτσα. Thank you. Ladies and gentlemen, it seems that Russia... Κυρίες και κύριοι, φαίνεται πως ε, η Ρωσία πέτυχε τον βασικό στόχο της και ο βασικός στόχος της ήταν να γίνει η Ουκρανία λιγότερο θελκτική από, ε, από τη Δύση. Και η Ρωσία συνεχίζει αυτή την προσπάθεια προκειμένου να μην καταστεί η Ουκρανία μέλος των δύο οργανισμών ο Πούτιν είχε πει ότι η Ουκρανία ποτέ δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δηλώνουν ότι οι πόρτες τους είναι ανοιχτές πάντα εάν φυσικά ο Ουκρανικός λαός το επιθυμεί. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διαφορετικά. Το παιχνίδι θα έχει κλείσει. Θα χάνουμε τον χρόνο μας και οι πολίτες μας ε, θα χάνουν και αυτοί τον δικό τους αλλά και εισοδήματα. Δεύτερον, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει μια νέα διακήρυξη δηλώνοντας σαφέστατα πως εάν ο Ουκρανικός λαός το θέλει, οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές προκειμένου να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ε, ενδεχομένω ε, ε, δυτικέ οργανώσεις. Δυστυχώς τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν κοινή θέση πάνω στο ζήτημα που μας απασχολεί για την τροσική εμπλοκή στην ουκρανική υπόθεση. Γι' αυτό λοιπόν οι κυρώσεις θα πρέπει να συνεχίσουν και ενδεχόμενα νέες κυρώσεις θα πρέπει να επιβληθούν στη Ρωσία διότι πρόκειται για θέμα τιμή, θέμα κόστους. Και για να κλείσω, τέλος αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να προωθήσει η Ουκρανία. Μιλάω για τα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Θα πρέπει να ενισχύσει περισσότερο τα σύνορα με την υπερνηστερία που δεν είναι αναγνωρισμένο έδαφος από τη Μολτανία, δηλαδή εξάγουν μέσω του λιμένα της Οδυσσού και δεν μιλάω τώρα για μεταρρυθμίσεις τα δικαιώματα των μειονοτήτων για να μπορούν να χρησιμοποιούν την μητρική γλώσσα και να διδάσκονται σε αυτή. Και τέλος να πω ότι τις τελευταίες ε, τοπικές εκλογές ε, το κόμμα που επιδοτήθηκε από την, Ευρωπα... από την ε, Μόσχα είχε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να κάνει το ίδιο με τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα της Μολδαβίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φραντζολίτσα. Παρακαλώ κύριε Τάνοκ σύντομα με σύντομη ερώτηση προς τον ε, κύριο Λατσμπερ και τον ε, πρέσβη. Αναφερθήκατε ότι αναφερθήκατε μάλλον στη συνεργασία ανάμεσα στην Γεωργία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Τι γίνεται με τον Γκουάμ, διότι εδώ δεν φεύγουμε τον ε, τροχό οργάνωση η βασίζεται σε μια συνθήκη και ο επεκτατισμός της Μόσχας πριν από μερικά χρόνια το κατέληψα αλλά και δεν έχω ακούσει, τίποτα σχετικά με την οργάνωση αυτή. Ευχαριστώ κύριο Καρατσαμπίλτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συναδελφοί μου ήδη είπαν αναλυτικά πως φοβερή είναι η κατάσταση σε αφορά την παραβίαση των ε, συμφωνίων του Μίνσκ. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση για την εξαιρετική εργασία που κάνουν εφαρμόζοντας τη Συμφωνία Σύνδεση. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να πω πω ε, πολλοί από μου προσπάθησαν να το πούν και λυπάμαι που χρειάζεται να το επαναλάβω. Εγώ ζητάμε από την ύπατη εκπρόσωπο τη ε, εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης τι κάνει σχετικά με τις παραβιάσεις π.χ. για τα εγκλήματα πολέμου, για τα ανθρωπιστικά εγκλήματα, τι γίνεται. Ξέρω ότι υπάρχουν 2.000 πρόσφυγες, 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, συγγνώμη. Σύμφωνα με την ΕΚΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει έλλειψη πρόσβασης ε, από πλευρά ΟΑΣΕ, υπάρχει ε, αδυναμία πρόσβασης των ανθρωπιστικών ε, αυτοκινητοπομπών. Πότε κυρία Μογκαρίνη θα θέσει το ζήτημα αυτό στην ατζέντα της, ε, του Συμβουλίου. Τι κάνετε για να εφαρμόσετε την ψήφισμα που το Κοινοβούλιο υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία, μάλλον δύο, δύο ε, ψηφίσματα. Τι θα κάνετε για να ενημερώσετε την δημόσια την κοινή γνώμη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το τι κάνει η, προπαγάνδα της Μόσχας. Εδώ συνάδελφος ήρθε σήμερα το πρωί και μας μίλησε για πόσα τάγκς και πόσες στρατικές δυνάμεις υπάρχουν στην Ουκρανία. Γιατί λοιπόν τα σιωπείτε όλα αυτά. Υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση η οποία είναι χειρότερη αυτή που είχαμε στο Σαράγεβο πριν από 20 χρόνια. Τότε λοιπόν η Ευρώπη δεν είχε μια εξωτερική κοινή πολιτική. Αλλά ο κόσμος κάθε μέρα έβγαινε στα μέσα ενημέρωση και έλεγε ότι είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Η Ευρώπη δεν ασχολείται. Τώρα έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Γιατί λοιπόν υπάρχει μόνο στα χαρτιά όταν αφορά στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Απέχω από το να θέσω το ερώτημά μου διότι τα είπε και ο κ. Κοράτσαμπίλ. Με κάλυψε κατά κάποιο τρόπο. Ο κ. Βίγκεν, επειδή πρόκειται να εγκαταλείψει σύντομα, παρακαλώ να ξεκινήσετε με τις απαντήσεις σας εξοχότατε. Well, I um, have listened carefully to you. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα λόγια σας κυρία Κορατσαμπίλντο. Νομίζω ότι δεν είναι απόλυτα ορθή η περιγραφή που κάνατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατηρήσει την συνοχή της και την ε, πολιτική της απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία. Και δεν νομίζω ότι είναι ίσονο σημασία το πείτε αυτό. Τώρα πολλοί από τους συναδελφούς ε, αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα. Αυτές οι κυρώσεις ε, διατηρήθηκαν ε, και πρόκειται στο εγγύς να ληφθούν νέες αποφάσεις. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτό γίνεται όχι με κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες αλλά με συνενέσεις. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και σύντομα θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Αλλά οι γραμμές έχουν δοθεί από το Συμβούλιο του Μαρτίου και αφορά στην πλήρη εφαρμογή της ε, συμφωνιών του Μίνσκ. Αυτό λοιπόν είναι το benchmark που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η κατάσταση στην ε, IDP είναι θέμα που μας απασχολεί. 1,3-1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες βρίσκονται στην Ουκρανία. Έχουμε χορηγήσει σημαντικά ποσά για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και όπως συχνά συμβαίνει κατά την περίοδο κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ε, μεγαλύτερος δωρητής, αλλά ε, υπάρχουν και άλλοι δωρητές που παρέχουν βοήθεια με αυτοκινητοπομπές και άλλους τρόπους ε, που φτάνουν σε περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου αλλά υπό τον έλεγχο άλλων και αυτή η ανθρωπιστική κρίση είναι απαραίτητη Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τις προσπάθειες ε, επικοινωνίας. Ε, εργαζόμαστε πάνω στο ζήτημα και θα υποβληθεί ένα πρόγραμμα δράσης προς το επόμενο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών Κυβερνήσεων. Ο Πρόεδρος σύντησε τι γίνεται με την ε, ομάδα Κόντι τέτοιες παρόμοιες ομάδες ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δύσκολες συναντήσεις ε, όπως την προηγούμενη φορά διότι ο Ρώσος εκπρόσωπος ε, αμφισβήτησε το όλο στήσιμο της ομάδας Κόντι διότι ζητούσε μια πλήρη συμμετοχή των οπαδών τους απόσκησης και αυτό Φυσικά δεν ε, βρήκε σύμφωνο ούτε όχι μόνο την Ουκρανία αλλά και τις άλλες, τα άλλα μέρη. Και στην τελευταία συνεδρίαση λοιπόν του μηχανισμού στο Παρίσι την περσμένη εβδομάδα ο Υφυπουργός τόνισε πως ε, υπάρχει ε, σημαντικός ρόλος που θα πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό, δεν θα... Αυτό αναφέρεται ρητά στις συμφωνίες του ΜΙΣΚ. Το ερώτημα του κ. Χάνικη που αφορά την ε, συμβουλευτική αποστολή της Ένωσης αυτό το οποίο μπορεί να γίνει τώρα για να κάνουμε καλύτερη χρήση αυτής της αποστολής είναι να συνεργαστούμε με τη δυνάμεις επιβολής του νόμου όχι μόνο στο Κίεβο αλλά και στις ε, διάφορες περιφέρειες. Αυτό άρχισε να υλοποιείται και θα υπάρξει μια επισκόπηση των ε, φθινόπωρο για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ενδεχόμενες ε, δραστηριότητε ε, κατάρτιση και εκπαίδευση. Το θέμα της αποκέντρωσης θα πρέπει να αποφασιστεί στο Κίεβο και να συνδεθεί με τις προσπάθειες ε, της ε, εφαρμογής της συμφωνία του Μίσκ. Όλοι γνωρίζουμε αυτήν την διτή πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Είναι αλληλεξαρτώμενες το Μίνσκ 2 έχει ενταφιαστεί, είπε η κυρία Γανιέτα. Και θα ήθελα, απαντώντας, να παραθέσω τον πρόσβη ότι δηλαδή το Μίνσκ είναι η μοναδική οδός για την ειρήνευση. Δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η σύραξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιούρης Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχάς, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Καταρχάς, εξοχότητες, κύριε και κύριοι, να σας ευχαριστήσω για την ε, υποστήριξη και την αλλαγή σας με την Ουκρανία. Βλέπω ότι το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της πλήρους εφαρμογής ε, τη συνθήκης του Μίνσκ και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται εν ώψη των δύο μεγάλων γεγονότων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Συμβούλιο ε, Εξωτερικών Υποθέσεων και το, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ελπίζω ότι θα ληφθούν υπόψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν τα ζητήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Αναμένουμε ότι τουλάχιστον θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ίδιες ε, κυρώσεις. Όχι όμως μόνο σε ό,τι αφορά τον Τόμπας, αλλά και σε ό,τι αφορά την Κρυμαία. Να σας υπενθυμίσω ότι οι κυρώσεις για την Κρυμαία θα εκπνεύσουν τον τρέχοντα μήνα. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσουν να ισχύουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Αδιάκοπα. Επίσης, ε, επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Φρόιντ για την πολύ καλή ερώτηση που θέσατε για τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Λυπάμαι, αλλά στην ομιλία μου δεν μπόρεσα να αναφερθώ σε όλες τις πτυχές της κατάστασης. Γιατί όντως η Ουκρανία αντιμετωπίζει δύο εχθρούς. Εξωτερική επίθεση από τη Ρωσική Ομοσπονδία και Α, κατά δεύτερον, εκ των έσω τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να διεξαγάγει. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι εκ παραλληλού είναι δύσκολο να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της τρέχουσα επίθεση, γιατί σκοπό της Ρωσικής Ομοσπονδία είναι να παρεμποδίσει και να αποσταθεροποιήσει ακριβώς ε, τη χώρα τι εσωτερικέ μεταρρυθμίσει, την οικονομική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση να μην επιτρέψει στην Ουκρανία να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύσκολο επίσης να επιβληθούν μεταρρυθμίσεις όταν κάθε μέρα αφαιρούνται μέσα 5 εκατομμύρια ε, δολάρια κάθε μέρα για τον πόλεμο στον Ντομπάς. έτσι όπως έχει η κατάσταση στο Ντόμπας και την Κρυμαία. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν πρέπει αυτό να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να μην γίνουν μεταρρυθμίσεις. Έχετε δίκιο όταν μιλάτε για την καταπολέμηση της διαφθοράς των ολιγοπολίων, των ολιγαρχιών, το οποίο ήδη δρομολογείται. Ε, επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Θα ήθελα να τονίσω και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις συζητήσεις που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Επίτροπος ε, για τα ανθρωπιστικά συστήματα προετοίμασε επίσκεψη στην Ουκρανία και 1η και 2η Ιουλίου αναμένουμε για τον κύριο Στυλιανίδη τον Επίτροπο με ένα σημαντικό πακέτο υποστηρίξης. Και σε ό,τι αφορά την αποστολή ΚΕΠΑ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να λεφτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια πραγματικά ορατή και διάκριτη υποστήριξη και παρότρινση για την εφαρμογή του Μίνσκ. Γι' αυτό που έθεσε ο κ. Τάνοκο ερώτημα. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σα. Και ξέρετε γιατί. Γιατί η Ουκρανία κατέχει την Προεδρία στο ΚΟΑ. Είμαστε σε διαδικασία εσωτερικών διαβουλεύσεων για την Γεωργία, το Αζερβαϊτζάν και τη Μολδαβία με σκοπό να δοθεί μια νέα πνοή στο έργο, στο πλαίσιο ΓΑΜ. Θα πρέπει λοιπόν να συζητηθεί αυτό επαρκώς. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι στο παρόν πλαίσιο θα πρέπει να δούμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση. Και πάλι κυρία Φωτίγκα, σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Αντρέη που συμμετέχετε στις διαβουλεύσεις και με τη βοήθειά σας θα κερδίσουμε. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρέσβη. Και να υπενθυμίσω στον κύριο Φραντζουλίτσα ότι την επόμενο μήνα θα επισκεφθεί την Μολδαβία και θα καταμετρήσει και θα αξιολογήσει τις συνέπειες της, ε, α, του εμπάρκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά δεύτερον, στα Ουκρανικά σύνορα, κατά δεύτερον ελπίζουμε να ακούσουμε την ανακοίνωση τις επισκέψεις όχι μόνο του Επιτρόπου Χαν, αλλά και της, ε, είπα, της εκπροσώπου κυρίας Μογκερίνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε ό,τι αφορά τους που χρειάζεται, προκειμένου να υπάρχει συνεχής παρουσία σε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα και σε μία από τις πιο σημαντικές περιοχές της ε, γειτονιάς μας. Ανδρέη, θα θέλεις να κάνεις καταλεκτικά σχόλια, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ να είσαι σύντομος. Ναι, να σας ευχαριστήσω μόνο. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ καλό α, το θέμα της συμφωνίας του Μίνσκ, γιατί θα γίνει και συζήτηση για τις νομικές μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση το, της διαφθοράς και προσβλέπουμε και στις 3 Ιουλίου την επισκέψη του πρόεδρου Σούλτς στην Ουκρανία για να υπογραφεί μνημόνιο στην εργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Ράντα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πρέσβευτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας στη σημερινή συνεδρίαση. Παρακαλώ μείνετε στην αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο της μέσας διάταξης απευθεία. Okay, Θα ξεκινήσουμε τώρα την ενημέρωση για την ε, ερενή σύνοδο της Κοινοβουλευτικής ε, Συνόδου του ΝΑΤΟ colleagues please please be seated those who, who would like Καθίστε παρακαλώ όσοι θέλετε να αποχωρήσετε παρακαλώ να το κάνετε σύντομα Uh, the uh, Η ε, αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρευρέθηκε τη διάρκεια τη συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Κίρτσος ήταν επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας, αντιπρόεδρος ε, της αντιπροσωπείας και θα ήθελα να του δώσω το λόγο για να μας ενημερώσει και μετά θα δώσουμε το λόγο στα υπόλοιπα μέλη. To, to, to contribute as well. Thank you very much. I would like to summarize some of... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνοψίσω κάποια από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα μετά τη συμμετοχή μου στην Ερηνή Κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πρώτον, οι περισσότεροι πολιτικοί και αναλυτές υπογράμμισαν ότι η Ρωσία θα εξακολουθήσει ε, να εφαρμόζει την επιθετική της πολιτική προς την Ουκρανία και θα ασκεί πιέσει στο ΝΑΤΟ και πολλά από τα μέλη της. Οι οικονομικές δυσκολίες στη Ρωσία και το πολιτικό κόστος που μπορεί να ενέχει για το καθεστώς αναγκάζει τον πρόεδρο Πούτιν και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του καθεστώτος να προσπαθήσουν να ενισχύσουν την εσωτερική του ε, θέση ακολουθώντας μια επιθετική εθνικιστική εξωτερική πολιτική. Φαίνεται ότι η οικονομία της Ουκρανίας πάει από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό δημιουργεί πολιτική και οικονομική αστάθεια που μπορεί να εξοπληθεί από του Ρώσου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ βεβαίω έχουν καθήκον να συνδράμουν την Ουκρανία για να υπερπηδήσει οικονομικέ και ε, άλλε δυσκολίε και να βοηθήσει στη σταθεροποίηση τη κατάσταση. Μια σταθερή και ενισχυμένη Ουκρανία είναι καλύτερη απάντηση στην επιθετική πολιτική της Ρωσίας. Εδώθηκε έμφαση στην υβριδική πολεμική μέθοδο που ακολουθεί ε, η Ρωσία και ότι χρειάζεται μία πιο ευέλικτη στρατηγική για να ε, καταπολεμήσουμε μεταξύ άλλων τη ρωσική προπαγάνδα. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα που ακολουθεί ο κύριος ε, Πούτιν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και δείχνει ότι επενδύει στη συνέχιση της συγκρούσης στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές. Από την άλλη, οι περισσότεροι αναλυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία δεν έχει την οικονομική και τεχνική, τεχνολογική μάλλον άνεση για να ολοκληρώσει αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα με βάση ε, τις ελπίδες και τους στόχους της. Περισσότερες συζητήσεις έγιναν και για την συμφωνία με το Ιράν, που θα είχε σημαντικά ωφέλη για τη διεθνή οικονομία. Ε, τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία έχουν παγώσει στο διεθνέ τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι ανάγονται μεταξύ 100 και 140 δι δολάρια. Ε, η οικονομική δυσκολία αλλά και το κράχ που θα μπορούσε να προκύψει σε περίπτωση που ε, αρθούν οι κυρώσεις δίνουν ε, πολλές δυνατότητες ό,τι αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες. Από την άλλη πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά ούτως ώστε το Ιράν να μην ε, αποκτήσει τελικά πυρηνικά όπλα. Οι κρίσεις σε χώρες όπως Συρία, Ιράκ και Λιβύη θα κλιμακωθούν εφόσον συνεχίζεται η αύξηση των ακραίων ε, Ισλαμιστών. Οι αποσταθεροποίησεις σε αυτές τις χώρες ε, επιδεινώνουν και επιτείνουν την μεταναστευτική ροή προς την Ευρώπη και καθιστά ακόμα πιο απαιτητική την εξέβριση λύσης στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να εξευρεθεί λύση από τους πολιτικούς και από τους αναλυτές και η ανάλυση που έγινε στην Ερηνή Σύνοδο είναι σωστή. Οι Ιρακινές δυνάμεις έχουν χάσει ακόμα περισσότερο έδαφος στους Ισλαμιστές και στη Λιβύη η ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται από την σεκταριστική πολιτική, βρίσκεται πλέον εκτός ελέγχου και ενισχύουν όλα αυτά τη μεταναστευτική ροή προς την Ευρώπη ε, σε κάνε φρεγουμένου. Υπάρχει και ένα ιστορικό μέτωπο με δεκάδες χιλιάδες νέους Ευρωπαίους που στρέφονται προς τους ακραίους Ισλαμιστές και ενδεχομένως να προσχωρούν και στις γραμμές τους. Πολλές χιλιάδες νέοι Ευρωπαίοι ήδη ε, συμμετέχουν στον ε, ένοπλο αγώνα στη Συρία και στο Ιράκ. Και αναφέρθηκε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μία περίπλοκη πολιτική για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε αυτά τα άτομα. Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να ε, εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις, τους, να αυξήσουν σταδιακά τις ε, δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα στο 2% του ΑΕΠ και να ε, εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα σε ό,τι αφορά και το σχέδιο ετοιμότητας του ΝΑΤΟ. Τέλος, ό,τι αφορά την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, η ε, δέσμευση προς την ε, πολιτική μας προς τη Σερβία, Ερζεγοβίνη, Βοσνία, ε, Φύρομ και Μαυροβούνιο, όλα αυτά επαναλήφθηκαν, όμως μόνο το Μαυροβούνιο θα λάβει πρόσκληση να προσχωρήσει στη συμμαχία πριν από το τέλος του 2015. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κίρτσο. Ο κύριος Βανόρντεν θέλει να πει κάτι. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ήταν πολύ υποδομητικές αυτές οι δύο-τρεις μέρες στη Βουδαπέστη. Εγώ παρακολούθησα κυρίως την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας της Κοινοβουλευτικής Συνόδου. Είχαμε λοιπόν μια πολύ επικαταματική ομιλία από τον ε, Αμερικανό στρατηγό, Νίκολσον, επικεφαλής ε, των ε, δυνάμεων στην Τουρκία. Και από τον Στίβεν Κάβινγκτον, στρατηγικός σύμβουλος και το σημείο εστίασης αφορούσε κυρίως τις νέες προκλήσεις στην Ανατολή και την κρίση στην Ουκρανία. Και η απάντηση που θα δοθεί από το ΝΑΤΟ με την ενίσχυση της ετοιμότητάς του. Πιο συγκεκριμένα βεβαίως Υπάρχει και κοινή task force. Μια ομάδα κρούσης 5.000 ε, στρατιωτών συν ενέργειες εξοπλισμός που μπορούν να τεθούν ε, σε κίνηση εντός 48 ώρων. Επομένω, πολύ σοβαρά τα εξετάζει αυτά τα ζητήματα το ΝΑΤΟ. Και αυτό ενισχύει τη θέση ότι το ΝΑΤΟ ε, είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μας και για την άμυνά μας και θα πρέπει καθόλου να αποδυναμωθεί. Υπήρξε συζήτηση και για αυτή την υβριδική πολεμική μέθοδο που ακολουθεί η Ρωσία. Και ιστορικά χρησιμοποιείται από τη Ρωσία και χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο για να πετύχει τους ε, πολιτικούς και άλλους στόχους της. Αναφερθήκαμε και ε, στο ζήτημα ISAF στο Αφγανιστάν. Πράγματι εξετάσαμε και αυτό το θέμα της ετοιμότητας και την ενίσχυση της διατελετικής σύνδεσης. Για τα κύρια σημεία που αναφέρθηκαν εκεί ήταν η πολιτική βούληση. Γιατί δεν πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα μόνο. Πρέπει να έχουμε και την πολιτική βούληση για τη στεναρή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ κύριε Βανόρντεν. Άλλα μέλη θέλουν να πάρουν το λόγο. Εάν όχι, να κλείσουμε τον κατάλογο, μάλλον ολοκληρώσουμε την εξέταση αυτού του σημείου. Παρακαλώ μείνετε στην αίθουσα. Σύντομα θα ξεκινήσει η δημόσια ακρόαση για την εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης από κοινού με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Παρακαλώ, μείνετε.